τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ομάδων του. Πρέπει επίσης με την επανάληψη των εργασιών μας να σας μεταφέρω ορισμένε θλιβερές ειδήσει. Ανακοινώσεις ε, για θανάτους τους ε, οποίους τώρα πληροφορούμαστε μετά τις διακοπές. Θεσνούμε τον συνάδελφο τον Ζήρι Χάβελ, έναν πάρα πολύ αγαπητό συνάδελφο που έχερε μεγάλη εκτίμηση. έναν εξαιρετικό πολιτικό, του οποίου οι εξαιρετικές γνώσεις ε, σημάδεψαν το έργο μας και το έργο της Επιτροπής ε, βιομηχανία και Προπολογισμού. Ήταν ένας παθιασμένος Ευρωπαίος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε και Μπορώ να πω πως αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην υπηρεσία των άλλων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης πενθεί την Edith Mastenbrook, της οποίας ο συγκλονιστικός θάνατος στην ηλικία των 37 ετών μας έθλιψε ιδιαίτερα. Αφήνει πίσω της ένα μικρό γιο, ο οποίος τώρα θα μεγαλώσει ορφανός. Θερνούμε επίση τον πρώην συνάδελφο Άλεξ Φάλκονερ και την Πάντι Λέιν, συναδέλφους οποίους ε, γνωρίσαμε σε προηγούμενες ε, θητείες και οι οποίοι επιπίεσαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι, ο Σβάλντο Παγιά και ο συναγωνιστής του Χάρολτ Σεπέρο, βραβευμένος ο κύριος ε, Σβάλντο Παγιά με βραβείο Ζαχάροφ, απεβίωσαν και οι δύο σε ένα ατύχημα στην Κούβα. Ο αγώνας ε, του Παγιά ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά στην Κούβα στον αγώνα τους για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίω αυτό ήταν το έργο της ζωής του Οσβαλτό Πάιες και γι' αυτό ακριβώς τον βραβεύσαμε το βραβείο Ζαχάροφ. και οπωσδήποτε θα τον θυμόμαστε. Θα ήθελα λοιπόν λόγω των προστιμήν των συναδέλφων οι οποίοι απεβίωσαν και του βραβημένου με βραβείο Ζαχάροφ να σας παρακαλώ να σηκωθείτε για ένα λεπτό Danke Ihnen. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι